Αγαπητοί συνάδελφοι, παραλαμβάνεται η συνεδρίαση από το σημείο που τη διακόψαμε χθε το απόγευμα και για σήμερα θεώρησα σκόπιμο πριν τις ευρωεκλογέ του επόμενου μήνα να οργανώσω μια τελευταία ανταλλαγή απόψεων για το δημοσιονομικό πλαίσιο του ίδιους πόρους για την περίοδο μετά το 2020. Και μάλιστα έχω το προνόμιο να συμπεριλαμβάνομαι στην διαπραγματευτική ομάδα με τους δύο συνεισηγητές για το δημοσιονομικό πλαίσιο Γιάνν Όλμπριχτ και Ιζαμπέλ Τομά και με τους δύο συνεισηγητές για τους ίδιους πόρους, τον Γιάννου Λεβαντόφσκι και τον Ζεγάρ Ντεπρέ. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να κάνω κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις αν μου επιτρέπετε εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Το Κοινοβούλιο εργάζεται ε, με ε, από κοινού για να δείξει πως είναι σοβαρό, υπεύθυνο, επικοδομητικό στο, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και θα ήθελα να σας αναφέρω την έγκριση δύο εκθέσεων πρωτοβουλία το Μάρτιο του 2018 για να δώσουν στοιχεία σε ό,τι αφορά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που Μας σε ένα ψήφισμα που με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς ε, μας επαναφέρει στα σωστά νούμερα, τα οποία η Κομισιόν δεν μας τα έδινε πάντοτε ε, σωστά. Και επίσης εγκρίναμε μια προσωρινή ενδιάμεση έκθεση τον Νοέμβριο με ρεαλιστικές, ποσοτικοποιημένες και αναλυτικές προτάσεις σαν ένα πρόγραμμα ε, με ένα έγγραφο αναφοράς το οποίο συνοδεύεται και από μέχρι προηγουμένου προσπάθεια συντονισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της ομάδας επαφής ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο του οποίο προεδρεύει ο ίδιος ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου κ. Σταγιάννη. Επίσης, με πρωτοβουλία των εισηγητών για το πολιετές και για τους ιδίους πόρους, οργανώθηκε μια σειρά συνεδριάσεων με τους εισηγητές για τα διάφορα τομεακά ζητήματα. Της ουσίας αυτό έχει επιτελεστεί ως έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν σταμάτησε όμω εδώ, αλλά τους τελευταίους μήνες η διαπραγματευτική ομάδα προσπάθησε να έχει όσο δυνατόν περισσότερο διάλογο με το Συμβούλιο στο πλαίσιο ενημερώσεων και απενημερώσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και στην συνεδρίαση ενός άτυπου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα το προηγούμενο μήνα στο Βουκουρέστι και είναι τακτική ανάγκη να ενταθούν με το νέο κοινοβούλιο οι επαφές αυτές. Εμείς επίσης προσπαθήσαμε γράφως να συμβάλλουμε στις συζητήσεις που δεν σε επίπεδο συμβουλίου. Διαδώσαμε κάποια σχόλια που είχαμε για τα διαπραγματευτικά κουτιά υπόψη των μελών του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όπως επίση και πιο συγκεκριμένα ημερωτικά δελτία για την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για όλες αυτές τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους τέσσερις συνεισηγητές, γιατί να με το Συμβούλιο από μόνο του ε, μονομερός ε, έχει καθυστερήσει ε, για τα τέλη 19 την έγκριση οποιασδήποτε τοποθέτηση για το πιδελταπή εμείς έχουμε προχωρήσει από την δική μας πλευρά με σταθερό ρυθμό, με συνέπεια και με πιστικό τρόπο και η διαπραγματευτική ομάδα που θα συγκροτηθεί ε, στη νέα θητεία θα πάρει τη σκητάλη και θα πρέπει να υπενθυμίσει και στο Συμβούλιο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι εξουσίες του Κοινοβουλίου στο, σε ό,τι δημοσιονομικό πλαίσιο δεν περιορίζονται στην απλή έγκριση στο τέλος της όλης διαδικασίας όταν δηλαδή θα πρέπει να, βάλουν, να δώσουν το πράσινο φως αυτό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ή αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πρόσχημα για να παρακαμφθούν οι προβλεπόμενες από τη συνθήκη νομοθετικές διαδικασίες. Επομένως, ε, στο πλαίσιο αυτής της ε, διαδικασίας θα πρέπει να γίνουν πραγματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για να είναι βέβαιο ότι θα δώσουμε εμείς την τελική μας έγκριση. Πρέπει επίσης να γίνουν σεβαστές οι εξουσίες συνάποβασης του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα προγράμματα και σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για το κράτος δικαίου. Παρά τις μερικές συμφωνίες οι οποίες έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες σε ορισμένα προγράμματα. Η βασική αρχή ε, αυτή παραμένει για όλες τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή τίποτα δεν θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί προτού συμφωνηθούν τα πάντα. Ήταν σαφές από πλευράς μας ε, αυτό. Θέλαμε να αποφύγουμε τη σχιζοφρένη, γι' αυτό θέλαμε να δούμε κοινώς ομού τις δαπάνες και, ε, και τα έσοδα και τους πόρους, που σημαίνει ότι στην πράξη θα πούμε όχι ως κοινοβούλιο αν δεν έχουμε πρόοδο και στο θέμα των ιδιών πόρων. Το πολιτές μεσομικό πλαίσιο και ήδη οι πόροι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Θα δώσω το λόγο στους εισηγητές ε, για να μας παρουσιάσουν το πώς έχει η κατάσταση. Για το πιδελταπικέ τους ίδιους πόρους. Τρεις είναι εδώ μαζί μας σήμερα το πρωί από τους τέσσερις. Ίσως ο Γιάνν Όλμπριχτ ε, θα μπορούσε να είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ενημερώσω απλά για το πώς έχει κατάσταση από την ε, πλευρά της ε, δικής τη δική μας, δηλαδή το πει κυρία Τωμά, δυστυχώς δεν είναι εδώ, αλλά θα προσπάσω εγώ να παρουσιάσω την κοινή μας θέση. Όλη η συζήτηση για το πολιτές οικονομικό πλαίσιο είναι ακριβώς αυτό που περιγράφατε, δηλαδή πηγαίνει προς ε, τρεις άξονες. Έχουμε το πρώτο σκέλος που είναι η συζήτηση για το πει και ο κανονισμός πει. Πρώτο στοιχείο αυτό που αφορά τα ποσά του προπολογισμού μηχανισμό, διάρθρωση, διάρκεια κτλ. Αυτό το πρώτο και βασικό στοιχείο. Και έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, έχουμε τη δική μας ε, θέση και αυτή εκφράστηκε στο πλαίσιο της ενδιάμεσης έκθεσης. Τώρα, για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάζει στην ενδιάμεση αυτή η έκθεση και κάποια νούμερα, αριθμητικά στοιχεία, τα με τα οποία προσπαθούμε να μεταφράσουμε την πρόταση της κόμισιο Σε συγκεκριμένα δηλαδή αριθμητικά στοιχεία. Η συζήτηση για το πι, για τον κανονισμό και το γενικό πλαίσιο, δεν έχει ολοκληρωθεί φυσικά, συνεχίζεται. Το συζητούν και ε, σε επίπεδο Συμβουλίου αλλά μόνο για ορισμένα σημεία, δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, γιατί υπάρχουν βαθιέ διαιρέσει ε, και υποκλήσει απόψεων μεταξύ των κρατών μελών, ιδίω ό,τι αφορά τα ποσά, αλλά και τη διάρθρωση και, για παράδειγμα, το ζήτημα τη ευελιξία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο για το πώς θα είναι τελικά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ο κανονισμός αυτός. Τι θα είναι, θα είναι αφετηρία ουσιαστικά για την ε, ε, ολοκλήρωση όλων των τομεακών κανονισμών για το ΠΔΕΛΤΑΠ. Όλα θα εξαρθούν από το ΠΔΕΛΤΑΠ επομένω. και όλοι εμείς περιμένουμε την κοινή θέση Συμβουλίου που θα πρέπει να ληφθεί με ομοφωνία και ανεπισήμως ε, με βάση το, το θεματολόγιο και την ε, ατζέντα των ηγετών θα πρέπει να την έχουν αποδεχθεί. Και εκεί διαβάζει κανείς αυτή την ατζέντα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει την πολιτική απόφαση πριν τα τέλη του έτους, ω τον Οκτώβριο, ως τον Νοέμβριο. Εν συνεχεία το Συμβούλιο και εν συνεχεία το Κοινοβούλιο που θα δώσει ε, και την έγκριση συμφωνή γνώμη, αν τη δώσει βέβαια. Δεύτερο άξονα. τα τομεακά προγράμματα που είναι απόρρια του πολιετούς. Σε αυτό το σκέλος ε, έχουμε δύο υποσκέλια αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι. Το ένα έχει να κάνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και το πώς διαπραγματεύονται μεταξύ τους για τους συγκεκριμένους κανονισμούς στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Στην ε, διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη. Για ορισμένα θέματα έχουμε καταλήξει. Για ορισμένα άλλα Έχουμε εν μέρη καταλήξει, για άλλα όμως δεν έχουμε καθόλου καταλήξει. Όπως ε, το CAP. Πήραμε όμως μια επιστολή. Την κοινωνική πολιτική δουλειά. Δηλαδή. Έχουμε πάρει μια επιστολή λοιπόν που λέει ότι έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο τριμερών διαλόγων μπορεί να καταγραφεί ως μερική συμφωνία όχι ως μερικό συμβιβασμό ή κάτι τέτοιο. Άρα, στον, ε, στην τελευταία σύνοδο του Απριλίου που θα ψηφίσουμε θα έχουμε την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για ορισμένες περιπτώσεις, για ορισμένα τομεακά προγράμματα θα έχουμε μερικές συμφωνίες. Αφού λάβουμε αυτή την επιστολή που ξεκαθαρίσει θέση του Συμβουλίου για το τι είναι μερική συμφωνία. Το τρίτο θέμα τώρα διαπραγματευτικά κουτιά και τομεακά προγράμματα. Αυτό έχει σχέση και με τη δεύτερη, ε, με το δεύτερο άξονα. Αλλά στο Συμβούλιο, πρώτα απ' όλα σα πω, τι κάνανε. Βάλανε σε αγκύλες ορισμένα ζητήματα. Δεν τα συζητάνε αυτά. Μόνο μεταξύ του τα συζητούν. Προετοιμάζοντα τη θέση του Συμβουλίου για τα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό. Πρώτον, Ακριβώ γιατί είναι δική μα αρμοδιότητα, στο οποίο στην απόφαση όπως πήγε ο πρόεδρό μας. Όμως το αφήνουν στου αρχηγού κρατών κυβερνήσεων που θα περιλάβουν αυτά ως απόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Αλλά πρόκειται για θέμα το οποίο θα έπρεπε να αποφασιστεί στο πλαίσιο τη διαδικασία συναπόφαση και δεν έχει καν συζητηθεί. Τι θα πρέπει λοιπόν να γίνει στο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα θα δεχτεί τα διαπραγματευτικά κοτιά που θα ψηφίσουμε στα τέλη του έτου. Αν παραλίλω δεν γίνουν αποδεκτά στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων με το Κοινοβούλιο, θα πρόκειται για μονομερή απόφαση του Συμβουλίου. Αν λοιπόν έλθει αυτή η απόφαση του Κοινοβούλιο, σήμερα νομίζω οι συγητές δηλαδή με τη σημερινή μας άποψη, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το κοινοβούλιο θα δώσει την έγκρισή του σε καμία περίπτωση, γιατί απαιτείται γι' αυτό τουλάχιστον στενή συνεργασία κατά την εκπόνηση της πρότασης. Και το κοινοβούλιο έχει αλλάξει, δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν πριν πέντε χρόνια. Και θα είναι και διαφορετικό μετά τις εκλογές. Είναι σημαντικό λοιπόν σήμερα, τα είπατε κι εσείς, σε ό,τι αφορά το κανονισμό για το ΠΔΕΛΤΑΠΗ. Δεν έχει ολοκληρωθεί τώρα, γιατί απαιτείται πολιτική τοποθέτηση σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Δεύτερον, οι τερμέρε διάλογοι συνεχίζονται, δεν μπορούν όμω να ολοκληρωθούν χωρί το ΠΔΕΛΤΑΠΗ. Και το διαπραγματευτικό κουτί είναι στη φάση της προετοιμασίας. Αν όμως δεν ληφθεί η άποψη του Κοινοβουλίου, θα υπάρχει μονομερής απόφαση. Η Ιζαμπέλ φαντάζομαι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι εμείς ως συνεισηγητές αυτό το οποίο αναμένουμε στο το τελικό στάδιο της όλης διαδικασίας είναι να υπάρξει εξέλιξη ε, είτε τέλη του έτου που είναι το πιο ε, αισιόδοξο σενάριο είτε τέλη του 2020 που είναι το λιγότερο είναι το πιο απεσιόδοξο σενάριο. Αν υπάρχει στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να περιμένουμε μάλλον το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτσι, όχι στο τέλο του τρέχοντος, το πρώτο εξάμεινο του επόμενου. Αυτό θέλουμε το αισιόδοξο σενάριο θα είναι το τέλο του 2020. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε. Γιάννα, Ποιο θέλει να πάρει το λόγο, κύριε Λεβαντόφσκι. Καλημέρα. Όσον αφορά τους ίδιους πόρους, ε, δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος μέχρι στιγμής. Τι απομένει τώρα για το Κοινοβούλιο και τους εισηγητές, τον Ζεράρ και εμένα, να επανεπιβεβαιώσουμε την θέση του Κοινοβουλίου, που είναι πιο φιλόδοξη από την αρχική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά την αιρεσιμότητά μας, ότι δεν θα γίνει συμφωνία για το PDP-ΔΠ αν δεν συμφωνήσουμε για τους ίδιους πόρους. 5 και 6 Απριλίου ε, θα έχουμε πρώτα απ' όλα στο Βουκουρέστι ε, την έκφραση της πρόθεσης να συζητήσουμε τους ίδιους πόρους. Ε, αυτή θα είναι μια πρώτη συζήτηση για τους ίδιους πόρους, πέραν από την δήλωση θέσεων υπέρ και κατά των νέων προσθήκων ε, στα πλευρά των εσόδων του προπολογισμού. Το ερώτημα είναι το κατά πόσο το κοινοβούλιο θα πρέπει να προσκληθεί. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει. Ε, συνίσταται μάλιστα ιδιαίτερο. Εγώ την Παρασκευή δεν μπορώ να βρίσκομαι στο Βουκουρέστι. Δεν ξέρω αν ο Τζέραρντ είναι διαθέσιμο για τη συνεδρίαση αυτή. Ακόμα δεν ξέρουμε αν μα έχουν καλέσει. Αν ο Τζέραρντ όμω είναι έτοιμο, καλό θα ήταν ε, να βρίσκεται εκεί στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας ώστε να συμβάλλει και αυτό στη συζήτηση μεταξύ των ηγετών ε, στην άτυπη αυτή συνεδρία της ΕΚΟΦΕΝ. Αυτά προς το παρόν. Θα μάθουμε την απάντηση. Ε, Ζεράρ, έχετε απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ τον Γιάννος για την πρόσκληση για το Βουκουρέστι, αλλά δυστυχώς έχω ήδη απαντήσει όταν με ρώτησαν για μένα είναι εντελώς αδύνατον. Δυστυχώς λυπάμαι. Δεν έχω πολλά να προσθέσω κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την κατάσταση των ιδιών πόρων και το θέμα αυτό, και εσεί ήσασταν στο Βουκουρέστι, συμμετείχατε στην τελευταία συνεδρίαση όπου αναφέρθηκε το πρόβλημα. Οπότε το μπαλάκι είναι στη δική σας πλευρά. Ε, έχετε μάθει κάτι θετικό από εκείνη τη συνεδρίαση. Στην φάση δεν έχω να πω παρά αυτά που υπενθυμίσατε εσείς και αυτά που μόλις είπε ο Γιάννης ότι για μας τα δύο ε, θέματα αυτά είναι αλληλένδετα. Τουλάχιστον για το παρόν κοινοβούλιο. Δεν ξέρω τι θα κάνει το επόμενο κοινοβούλιο. Διότι η σύνθεσή του δυστυχώς θα είναι λίγο διαφορετική μετά από τις επόμενες εκλογές. Ε, Εύχομαι η ψήφο των πολιτών να ακολουθεί την καλή λογική και όχι την κακή. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Υπάρχει ένα στοιχείο νέο το οποίο ενδεχομένω θα ε, επισέλθει. Πλησιάζει ο χρόνος. Μάλιστα το τι θα γίνει με το Brexit. Σε περίπτωση σκληρού Brexit τίνω να πιστεύω ότι οι διπόροι θα γίνουν πιο απαραίτητοι. Ε, εγώ θεωρώ αυτό ότι μπορεί οι μπορεί να γίνουν πιο σημαντικοί από ποτέ διότι θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε σημαντικά τις ε, εθνικές συμμετοχές ε, στο αντίθετο σενάριο. Οπότε πρέπει να σας πω δεν θέλω να γίνει σκληρό Brexit για να έχουμε δύο σπόρους, αλλά πιστεύω ότι θα επηρεάσει σημαντικά τη συζήτηση που θα γίνει σε επίπεδο Συμβουλίου. Αλλά στην παρούσα φάση, όπω είπε ο Γιάννου και όπω επαναλάβετε κι εσεί, ένα έχουμε να πούμε ότι τα δύο αυτά θέματα είναι αλληλένδετα. Χωρίς, δεν θα υπάρξει συμφωνία του Κοινοβουλίου εάν δεν σημειωθεί πρόοδο στον τομέα των ιδιών πόρων. Eh bien, Μάλιστα, κύριε Σιγητά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε άλλα επιχειρήματα. Πέραν τη ε, Brexit χωρίς συμφωνία. η πιθανότητα να παραμείνει ακόμα στο κοινοβούλιο το Ηνωμένο Βασίλειο για κάποιους μήνες ε, διαγράφεται πιο καθαρά. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε κάποια σχετική εκστρατεία. Θα πρέπει να μας απασχολήσει στις επόμενες μέρες το θέμα. Προηγουμένως, ο, ε, ε, μου έλεγε ο διευθυντής της DG Badge ότι έχει στείλει ήδη την επιταγή του Ηνωμένου Βασίλειο για τον Απρίλιο. Ναι. Ε. Τέλο πάντων, αφού αναφερόμαστε στο ΠΔΠ και του ίδιου πόρου, δίνω το λόγο τώρα στου ο ηγητέ, τον κύριο Φερνάντε. Όχι. Η κυρία. Κατία παρακαλώ. Όχι, ο κύριο Κέλμελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα για τις ε, τεχνικές λεπτομέρειες νομίζω δεν έχω να προσθέσω κάτι, να κάνω κάποια παρατήρηση. Ο Ζεράρ, ο φίλος μου, επιβεβαίωσε αυτά που σκέφτομαι και εγώ. Και τα είπε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζει δηλαδή οι πολίτε να έχουν ε, λάβει τη σωστή απόφαση, είπε. Εγώ νομίζω πω οι πολίτε πάντα λαμβάνουν τι σωστέ αποφάσει. Α, και εμείς οφείλουμε να δεχτούμε την απόφαση των πολιτών, ακόμα και αν δεν μας αρέσει. Εγώ το δέχομαι. Και για όσους ε, δεν συμφωνούν, να σας θυμίσω το βιβλίο που ε, έχει ως ήρωα έναν βασιλιά που δεν θέλει το λαό του και αποφασίζει να βρει έναν άλλο λαό να κυβερνήσει δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο χωρίς να σημειωθεί πρόοδος για τους ίδιους πόρους. Τι σημαίνει αυτό, ότι μέχρι σήμερα έχουμε μία βάση με ίδιους πόρους και υπάρχουν προβλήματα, δεν τους θέλουμε. Μετά τον Brexit όμως, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, τι θα κάνουμε. Θα λέμε δεν έχουμε προπολογισμό. Νομίζω πως πρέπει να ξανασκεφτούμε λίγο αυτή τη θέση και εάν υπάρχουν εύστοχα επιχειρήματα για τους ίδιους πόρους να τα δεχτούμε. Εάν δεν μας πείσουν τότε δεν θα μπορέσει να σημειωθεί πρόοδο στο θέμα των ίδιων πόρων. Νομίζω πως είναι ένα ε, θέμα αρχής. Τι θα κάνουμε αν δεν έχουμε πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ότι θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος άλλος δεν θέλει το λόγο. Κύριε Βανκά. Hm. Ευχαριστώ πολύ. Οι ήδη πόροι σίγουρα είναι πολύ σημαντική και εμείς πρέπει να τηρήσουμε τις ε, δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συνθήκες και όχι μόνο λόγω του Brexit. Όταν υπήρχε η ομάδα Μόντι, είχαμε πολύ καλή εκπροσώπηση και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ε, προετοιμασία για την πρόταση με τους ε, ίδιους πόρου, είχαμε κοιτάξει το θέμα από κάθε πιθανή οπτική γωνία και στο τέλος το πόρου ήταν ομόφωνο. Μόνο ίσως ε, ένα μέλος της ομάδας είχε άλλη άποψη. Τώρα βέβαια θέλω μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το γιατί η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν έχουν δεχτεί κάποια στοιχεία της έκθεσης Μόντι. Το μόνο επιχείρημα που έχω ακούσει είναι ότι δεν μπορούν να δεχτούν την φορολόγηση άνθρακα, για παράδειγμα. Αλλά θα ήθελα να μάθω τα επιχειρήματα. Ο φόρος άνθρακα είναι ε, κάτι που μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς στόχους. Πρώτον, να αναγκάσει τις τρίτες χώρες να έχουν πιο αποτελεσματική παραγωγή αγαθών και να επιτύχουν τους ε, στόχους για την καταπολέμηση της ε, κλιματικής αλλαγής. Να αυξηθεί λοιπόν η ανταγωνιστικότητα και να αναγκάσει τις χώρες ε, του τρίτου κόσμου να αλλάξουν στάση και να αποφέρει έσοδα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Επιτροπή γιατί αυτά τα στοιχεία έχουν μείνει εκτός το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ήταν πάρα πολύ καλό, θεωρώ. Όμω, όταν κάτι δεν συμπεριλαμβάνεται ε, και μένει απ' έξω, νομίζω θα πρέπει να αιτιολογείται. Και αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμή. Ευχαριστώ. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιο άλλο θα ήθελε να πάρει το λόγο για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και του ίδιου πόρου. Κύριε Φερνάνδε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τέσσερις συνεισηγητές και τις πολιτικές ομάδες ε, που εργάστηκαν για το θέμα αυτό. Έγινε πολύ καλή δουλειά. ώστε να υπάρξει μια καλή συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογέ. Και περιμέναμε το Συμβούλιο το οποίο ακόμα δεν έχει λάβει θέση. Τι μπορεί τώρα να συμβεί στο μέλλον. Το Συμβούλιο δεν ασχολείται με τις εργασίες του Κοινοβουλίου και αποφασίζει μόνο του και υποβάλλει την πρότασή του σαν κάτι που τετελεσμένο, το οποίο ή το δέχεσαι ή το όχι. Και να παίξει ένα χάρτη εναντίον του Κοινοβουλίου λέγοντας ότι αν το Κοινοβούλιο δεν δώσει την έγκρισή του δεν θα έχουμε πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έγκαιρα για το 2021. Θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό τέτοιο παιχνίδι, τέτοια πίεση μπορεί να ασκήσει και να παίξει το Συμβούλιο. Και εμείς δεν θέλουμε να βρεθούμε πρωτετελεσμένων. Έχουμε κάνει τη δουλειά μας έγκαιρα και είναι και καλή δουλειά. Και τώρα το Συμβούλιο, όπως είπαν οι εισηγητές, θα πρέπει να δείξει σεβασμό προς τους πολίτες. Δηλαδή, θα πρέπει να έρθει να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο. Συγγνώμη. Στον τομέα των ιδιών πόρων, επίση θα πρέπει να είναι τα πράγματα σαφή για μας οι ίδιοι πόροι. Δεν συνεπάγονται μόνο μείωση και υποκατάσταση, αντικατάσταση ε, εθνικών δαπανών και προϋπολογισμών. Τι εννοώ, τα έσοδα των ιδίων πόρων θέλουμε να συμβάλλουν σε αύξηση του προϋπολογισμού στο επίπεδο που ε, υπερασπίζεται το Κοινοβούλιο και όχι μόνο για να μειωθούν οι συμμετοχές ε, των εθνικών προϋπολογισμών. Αυτό πιστεύω είναι η πρόθεση του Συμβουλίου. Αντικατάσταση και να διατηρηθεί ο προπολογισμό στο ίδιο επίπεδο. Ζητάμε 1,3 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δεν είναι κάτι εξωφρενικό. Ούτω ώστε να τηρούμε και τι προτεραιότητε του Συμβουλίου. Ούτω ώστε να καλυφθούν τα ποσά που χρειαζόμαστε για την πολιτική συνοχή, στην αγροτική πολιτική, την έρευνα, το Εράσμους, τι νέε προτεραιότητε. 1,3 δεν είναι κάτι εξωφρενικό και είναι μια καλή μεθοδολογία αυτή, η μεθοδολογία της προσθήκης. Δηλαδή ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, ε, ε, του αθρίσματο, συγγνώμη, και τη πρόσθεση του αθρίσματο. Μετράμε τι προτεραιότητε, τι αθρίζουμε και βλέπουμε τι χρειαζόμαστε. Το 1,3 δεν είναι εξωφρενικό. Σε πολλέ χώρε το 1,0 ε, το ακαθάριστο εθνικού προϊόντο λένε να δώσουμε. Κρατάμε ό,τι είχε δώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, ίσω η γραμμή ε, για τα δημοσιονομικά της Ευρωζώνης να συμπεριληφθεί και αυτή και μετά να διαιρέσουμε αναπροτεραιότητα. Έτσι δεν δείχνουμε σεβασμό προς τους πολίτες, ούτε ενδυναμώνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω τους τέσσερις συζητητές για την άριστη προσπάθειά τους. Ευχαριστούμε. Ποιος άλλος. peut Ίσως να καταφέρουμε να βρούμε 12-14 δισεκατομμύρια πόρων, ε? διότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, euh, Λίγο πρόωρο, ε εντάξει, να ε, κάνουμε προβλέψεις για τους πόρους αυτούς. Κοιτάξτε, ένα στοιχείο εμένα με έφερε σε δύσκολη θέση. Δεν έγιναν συζητήσεις εκ των προτέρων για να ξέρουμε για ποια Ευρώπη μιλάμε. Συζητάμε έναν προπολογισμό για την περίοδο 2021-2027. Αλλά τι μορφή θα έχει η Ευρώπη το 2027 θα είναι μια παγκόσμια δύναμη. Αυτό θέλουμε. Αν θέλουμε να την καταστήσουμε παγκόσμια δύναμη, που να μην είναι υποταγμένη στην Κίνα ή σε άλλες χώρες, διότι δεν καταφέρνουμε να ισοσκελίσουμε τους δικούς μας εθνικούς προϋπολογισμούς ενίοτε, αυτό τι σημαίνει από δημοσιονομική άποψη. η αρχική κρατών και κυβερνήσεων λοιπόν τι θα αποφασίσουν δεν ξέρω. Εγώ με τον κύριο Αλμπρεχτ όταν συναντηθήκαμε με τους υπουργούς, ε, τους υφυπουργούς ε, και κάποιους ε, επικεφαλής διοικήσεων σχηματίσαμε την εντύπωση ότι λένε αυτά που λένε εδώ και μήνες στις κυβερνήσεις τους χωρίς πραγματικά να έχει προγραμματιστεί οτιδήποτε, να έχει σχεδιαστεί οτιδήποτε. Σαν να μην έχει ξεκινήσει καν η διαπραγμάτευση. Μα έδωσαν την εντύπωση ότι αναμένουν κάποια διαιτησία από τους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων σε κάποια σύνοδο κορυφής. Αυτό που φοβάμαι δηλαδή είναι ότι ξαφνικά θα συμφωνήσουν κάτι χωρίς απαραίτητα να λάβουν υπόψη τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Δεν ήμουν εδώ το 2013, αλλά θεωρώ ότι ε, αυτό που είχε επιτευχθεί τότε ήταν άνευ προηγουμένου. Και ίσως ε, θα πρέπει αυτό να αντιληφθούμε κάποια στιγμή, ότι ε, να αντιληφθεί μάλλον το Συμβούλιο, να σταματήσει να θεωρεί ότι σε θέματα δημοσιονομικά το κοινοβούλιο εξαρτάται από τις αποφάσεις των, ε, και δέχεται τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Αυτό εγώ ε, αισθάνθηκα μερικές φορές ε, στις αιτήσεις διαδικασίες συνδιαλλαγής. Ξεκινάμε μία διαπραγμάτευση όλο φιλόδοξη, πολύ φιλόδοξη, λέγοντας διάφορα μεγαλόσχημα λόγια και μετά όταν φτάνουμε στην τελευταία φάση η αποφασιστικότητα κάμπτεται. Και κάθε φορά γίνεται το ίδιο. Κάποια στιγμή λοιπόν τα πράγματα θα πρέπει να έχουν άλλη έκβαση. Να υπάρξει και κάποια αντιπαράθεση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να καταβάλουμε για να έχουμε σεβασμό, για να λαμβάνετε υπόψη η απόψή μας. Και μετά για τους ίδιους πόρους, ε, και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Όταν λέμε ότι οι διπόροι θα αυξήσουν τη φορολογική επιβάρυνση για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, ε, δεν είναι και ο καλύτερο τρόπο για να προωθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγοντα, ε, ακόμη και αν λέμε ότι οι διπόροι θα ληφθούν από φόρου που δεν πληρώνονται, δεν καταβάλλονται απευθεία από του Ευρωπαίου πολίτε. Αλλά παρόλα αυτά θα μα έρθει μπούμεραγκ. Όταν ε, ζητάμε από τι τράπεζε να πληρώσουν φόρου, τελικά όσοι παίρνουν δάνεια, οι δανειολήπτες ε, καταβάλουν τους φόρους αυτούς που έχουν να καταβάλουν οι τράπεζες. Ε, και αν είναι να πάρουμε από τα ακουστικά μέσα ας πούμε κάποιους φόρους αυτοί θα ζητήσουν από τους διαφημιστέ. Ε, οι διαφημιστέ θα ζητήσουν από κάποιου βιομηχανου οι οποίοι μεταφέρουν τι παραγωγέ στην Ασία και τελικά θα την πληρώσουν οι καταναλωτές Οπότε, ας μην ε, ε, συζητάμε για νέους πόρους, γιατί δεν ε, επισέρχονται στην εξίσωση. Όταν μιλάμε για ίδιους πόρους, ουσιαστικά είναι για λαφρύνουμε την δίκαιη επιστροφή, αυτή την τυραννία, όπου κάθε κράτος συγκρίνει ό,τι λαμβάνει από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό υπό τη μορφή Ταμείων Συνοχή ή Κοινή Γεωργική Πολιτική και να το αντιπαραβάλει αυτό με τη δική του συμβολή στον προπολογισμό, με δύο κατηγορίε κρατών, του ε, καθαρού ε, ε, συμβάλλοντε και του. τους καθαρούς εισφορείς και τους καθαρούς δικαιούχους. Οπότε αυτό στις 2 Ιουλίου θα συνεχιστεί αυτό που είχαν κάνει πάρα πολύ ωραία οι συγητές μας και εκεί θα έχουμε μια δοκιμασία που το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα η αναγνώριση του Κοινοβουλίου ως ένας θεσμού που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως η Κομισιόν μέσω του Γενικού Διευθυντή Κοκμάν θα μπορούσε να μας διαφωτίσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να διαφωτίσω τη συζήτηση. ούτως ή άλλως είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα έχει συζήτηση μέχρι τώρα. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι φυσικά και δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι σαφές ότι το Συμβούλιο ε, προχωρά με το δικό του τρόπο και κατανοώ απολύτω και τις ανησυχίες και τα ερωτηματικά σας. Όμως ακούγεται η άποψή σας. Οι υπουργοί γνωρίζουν πολύ καλά πως ήδη ίδιοι πόροι είναι ένα πολύ σημαντικό για το κοινοβούλιο ζήτημα και ότι τελικά η θέση σας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κατά την άποψή μου λοιπόν, η μόνη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω είναι να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε πολύ καλά. Δηλαδή να είστε τεχνικώς προετοιμασμένοι, ήσασταν οι πρώτοι μεταξύ των θεσμικών οργάνων που καταθέσετε συγκεκριμένε αναλυτικέ ποσοτικοποιημένες προτάσεις ουσιαστικά αναγκάζεται το Συμβούλιο να δραστηριοποιηθεί, να δεσμευτεί, συμμετέχετε στις, οργανώσεις, ε, στις συνεδριάσεις που οργανώνονται και σίγουρα πρόκειται για μια διαπραγμάτευση και υπάρχει ένα άλλο θεσμικό όργανο που ακολουθεί μια διαφορετική λογική. Εγώ δεν θα κάνω σχόλια, δεν είναι η δουλειά μου. Όμως και εσείς ακολουθείτε τη δική σας λογική και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι μια λογική η οποία έχει ε, λογική, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεύτερον, η συζήτηση για τους ίδιους πόρους. Ε, είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή. Και όλα τα επιχειρήματα του Προέδρου για το πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει πολύ σημαντική αύξηση των δυο πόρων. Είναι πολύ εύστοχα και βάσιμα. Αλλά και η θέση σας, όπως την έχετε εκφράσει, είναι σημαντική. Δηλαδή ότι απαιτείται κάποια μεταρρύθμιση του του συστήματος παρόλα αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ, παρά τις δυσκολίες επίπεδο Συμβουλίου, οι συνάδελφοι του Συμβουλίου ακούν. Τίνουν ευήκον ούση κομισιών, προασπίσει προτάσεις της. Ε, έχουμε προτείνει κάποια έως νεοτερισμούς. Και στη τελική ανάλυση εδώ είναι ένα σημείο δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το λάβει υπόψη στον προβληματισμό του το Υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο που το Κοινοβούλιο πάντοτε επηρέαζε σημαντικά το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Μιλάω για την ευελιξία. Οι εκπρόσωποι σα στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στο Βουκουρέστι εξέφρασαν τις απόψει τους και τα επιχείρηματά του και μπορώ να σα επιβεβαιώσω ότι έγινε ακουστή η άποψη αυτή. Και αυτό είναι σημαντικό για τη λειτουργία του προπολογισμού, για την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σας ε, συμβουλεύω λοιπόν να το έχετε αυτό κατά νου και γνωρίζετε πολύ καλά ότι το κοινοβούλιο σας είναι αυτό το οποίο στην ενδιάμεση αξιολόγηση κατάφερε να καινοτομήσει στον τομέα αυτό. Όλα αυτά γιατί σας τα λέω, για να σας ε, καταδείξω τη σημασία του ρόλου σα. Είναι ένας έντιμος τη Κομισιόν και από αυτό το ρόλο συνεργάστηκε με εσά και με το Συμβούλιο. Και ελπίζουμε πω η αφοσίωση, η προσήλωση, ο ζήλο σα θα παραμείνουν ε, ανέπαφοι και του επόμενου μήνε και όταν θα αλλάξει τον Ιούλιο η σύνθεση του Κοινοβουλίου. Γιατί νομίζω ότι σας χρειάζεται η Ευρώπη για να φτάσει σε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Γραμματέα. Μας χαϊδεύουν τα αυτιά αυτά που είπατε, είναι ενθαρρυντικά λόγια και σίγουρα θα τονώσουν και την αυτοπεποίθησή μας. Όσοι συνάδελφοι λοιπόν είναι εδώ και στην προσεχή θητεία, έχουν βλέπουμε αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη των συναδέλφων. Ήδη εξασφαλισμένοι από τώρα και στην ιατρική επίσης βλέπουμε ότι μπορεί να είναι η πρόοδος μέτρια, αλλά το σημαντικό είναι να πηγαίνει σωστή κατεύθυνση. Και αυτό έχουμε πετύχει, αυτό έχει κινητοποιηθεί. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν στη μέση της διαδρομής. Επιτροπή Προϋπολογισμών με την εμπειρία της σίγουρα θα επανεπιβεβαιωθεί στο ρόλο της, ε, θα παρακινηθεί λοιπόν να συνεχίσει τις εργασίες της και στην επόμενη και αυτό προνείστε μόνο καλά για την Ένωση και το μέλλον της. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συνεισηγητές, αρχίζω αυτή τη φορά από τον εισηγητή για τους ιδίους πόρους, αν μπορεί να μιλήσετε κανένα δεκάλεπτο ακόμα, καλά θα ήταν. Γιατί στις 10 έχουμε το επόμενο θέμα μας μόνο. Κύριο κύριος Τεπρέ. Κύριε Τεπρέ, κύριε Πρόεδρε, θα μιλάω αργά, ώστε να καταλάβουν όλοι πολύ καλά. Μάλιστα, λοιπόν, ανταλλάξαμε επένους και εγκόμια, ε, πολύ δικαιολογημένα νομίζω, γιατί πράγματι εργαστήκαμε με σοβαρότητα και πράγματι δεν το 2013 και ε, μάλλον ήμουν το 2013 και κάναμε σοβαρή δουλειά. Νομίζω από το τι έγινε παλαιότερα. Άκουσα πολύ προσεκτικά το Γενικό Διευθυντή. Ε, δεν έχει όμως υποθεί κάτι. Θέλω να το πω. Μπορεί και να μην είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο της πρότασης, όμως η πρόταση της Κομισιόν για τη διαπραγμάτευση ήταν μια καλή βάση συζήτησης για εμάς. Ε, έκανε κάτι που το είχαμε ζητήσει και το λέω στο Γενικό Γραμματέα προέβλεψε δύο πτυχές αυτές που είναι σημαντικές για εμάς ε, άμυνα και ήδη πόροι ε, μάλλον δαπάνες και ήδη πόροι euh, έτσι καταφέραμε και εμείς να εργαστούμε ποιοτικά. Είπε κάτι ο συνάδελφος Κέλμελ. Θέλω να το τονίσω οι νέοι διπόροι, το είπε και ο Ζωζέ. Δεν είναι μόνο για να καλυφθεί η τρύπα από την ενδεχομένη αποχώρηση των Βρετάνων και τιμέ των κονδυλίων. Θα χρειαστούν οι διπόροι νέοι ούτω ή Υπάρχει όμω ένα σημαντικό στοιχείο το κοινοβούλιο. Αν έχει ίδιου πόρου σε σχέση και με τη δική μας πρόταση. Δηλαδή, από τη στιγμή που λέμε ότι σε έναν τομέα, παραδείγματος χάρη, φόρος επί των εταιριών εφόσον θα έχει ενοποιηθεί η κοινή φορολογική βάση και θέλουμε ένα μέρος αυτού του προϊόντος να πηγαίνει στον προϋπολογισμό. Υπάρχει ε, ένα αυτόματο μηχανικό στοιχείο. Δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να επαναδιαπραγματευόμαστε τη χρηματοδότηση του συνόλου του προπολογισμού με τα κράτη. Δηλαδή θα υπάρχει ένα άλλο και πιο σημαντικό κομμάτι το οποίο μηχανικά αυτόματα θα προκύπτει από την ε, συμπερίληψη ορισμένων φόρων ε, με το σύστημα ΦΠΑ, το νέο, όπως προβλέπεται στη γόντια της Κομισιόν. Έχουμε αυτόματα αύξηση της απόδοσης. Αν έχουμε αύριο το ίδιο με τον εταιρικό φόρο ή με ένα μέρος ε, του φόρου από το ETS, την εμπορία εκπομπών. Έτσι τροφοδοτείται ο προπολογισμό και δεν χρειάζεται πλέον να λαμβάνονται αποφάσει και να υπάρχει διαπραγμάτευση κάθε χρόνο για το κάθε σεντ. Και αυτό είναι ενδιαφέρον κύριε Κέλμελ. Μεταξύ άλλων και αυτό είναι ενδιαφέρον. Υπάρχουν και άλλα ότι με την αποχώρηση των Βρετανών ε, επίσης θα επηρεαστούν ε, αυτόματα οι εκπτώσεις, οι επιστροφές που δεν δικαιολογούνται πλέον. Άρα θα γίνουν κάποια πράγματα, θα χρειαστεί να γίνουν κάποια πράγματα και η αναδιαπραγμάτευση των δύο πόρων είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δεν είναι ένα απλό παζάριμα μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών για τον τρόπο με τον οποίο θα αντισταθμιστεί το ένα ή το άλλο. Και η Ιζαμπέλ και εγώ πάντοτε, μάλλον ο Γιάννη και εγώ πάντοτε θέλαμε να έχουμε ένα καλάθι για να υπάρχει εξισορρόπηση και όχι δυσανάλογη εκπροσώπηση, συμμετοχή των κρατών παρά την οικονομική τους κατάσταση. Μίλησα κανένα πεντάλεπτο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο όμως, Πρόεδρε. Έτσι είναι η κατάσταση. Και δεν θα έχουμε το προνόμιο να σας έχουμε πρόεδρο και στην επόμενη θητεία. Θα πω ότι θα έχω την τύχη και την ε, ατυχία ή μάλλον δεν θα έχω την την ατυχία, δεν ξέρω αν είναι πρωτό, προνόμιο ε, στην επόμενη θητεία. Πάντω θέλω να πω από τώρα ότι ήταν πολύ μεγάλη χαρά που ήμουν εδώ, γιατί εργαστήκαμε πολύ δουλειά στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ. Θα δούμε 5 Ιουνίου τι θα γίνει. Ε? Σε τέσσερα λεπτά πρέπει να πάω για ψηφοφορία στην Ήτρε. Και έχω μόνο δύο λεπτά τώρα για να σας πω γιατί ο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και για τους ίδιους πόρους. Μετά από τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, τι έγινε, ποια ήταν η προοπτική το 2006, ήταν η τελευταία φορά που καταφέραμε, εγώ ήμουν στην Επιτροπή Κόμη, να αυξήσουμε τον προπολογισμό κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό έγινε την τελευταία φορά. Μια πραγματική αύξηση, όχι πολύ μεγάλη, αλλά αύξηση παρόλα αυτά μετά από διαπραγματεύσει. Αυτό ήταν για το πολιτε δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 και στον τελευταίο γύρο υπό την πίεση του κ. Κάμερον υπήρχε απελπιστική ανάγκη να δοθεί περισσότερη ευελιξία στον προπολογισμό. Αφορούσε το ζήτημα μόνο την ευελιξία, όχι τι αυξήσει και ε, είχαμε και την ομάδα Μόντι για τους ίδιους πόρους τι θα είχε γίνει χωρίς τον κύριο Κάμερον, ποια θα ήταν η έκβαση των διαπραγματεύσεων, χωρίς την πίεση ε, και τη μεγάλη αντοχή, που, ε, τη μεγάλη αντίσταση που υπήρξε στην πρόοδο, δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι σαφές, ο λόγος για τις προϋποθέσεις αυτές είναι διότι είναι πολύ ισχυρότερη θέση μας όσον αφορά τις δαπάνες από ό,τι για τα έσοδα Οπότε επικαιροποιήσαμε το φάκελο των, νέων πόρων, των ιδιών πόρων για τι διαπραγματεύσει. Αυτό είναι ο πραγματικό λόγος. Ε, και μιλάμε και για μειώσεις ε, από το ακαθαρίστον χώριο προϊόν. Αυτά. Ευχαριστούμε. Στον πρώτο γύρο έγιναν λοιπόν οι επίσημες δηλώσεις και στον δεύτερο γύρο, όπως καταλαβαίνω, λέμε αυτό πραγματικά πιστεύουμε. Θεωρώ πως ε, δύο στοιχεία είναι σημαντικά εδώ. Πρώτα, το Brexit. Αν κάτι πάει στραβά τις επόμενες μέρες, τότε η συζήτηση θα είναι τελείως διαφορετική. Διότι στην ουσία αυτό που συζητάμε είναι ο προπολογισμό μετά το 2020. Φανταστείτε να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα-δύο χρόνια ακόμα το πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχει τελείω διαφορετική μορφή με όλες τις εκτόσεις ε, που αυτό συνεπάγεται κτλ. Οπότε είναι μια τελείως ε, διαφορετική εναλλακτική. Έπειτα, Αυτό που προσπάθησα να εξηγήσω και κατά την ε, τελευταία πενημέρωση με τη Ρουμανική Προεδρία είναι ότι οι υπουργοί της Προεδρίας συνειδητοποίησαν ότι το Κοινοβούλιο έχει μάθει πολλά και διαφέρει από όπως ήταν πριν από πέντε χρόνια. Αυτό γιατί πρώτον ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο και δεύτερον έχουμε και την εμπειρία. Δηλαδή λέμε ή το παίρνεις ή τα αφήνει. Το Συμβούλιο όταν δεν δέχεται κάτι λέει τέρμα. Όμως το 2020 είναι ένα έτος μετά τις ευρωεκλογέ και όχι πριν τις ευρωεκλογέ και αυτό αλλάζει πολλά ως προς τη στάση του Κοινοβουλίου. Ε, μπορεί δηλαδή να ε, εμπεριέχει πρόταση μεγαλύτερο ρίσκο. Έπειτα, ε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια κοινή θέση εντός του Κοινοβουλίου. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Όλοι προερχόμαστε από διαφορετικές θέσεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μία κοινή, κοινά αποδεκτή θέση από όλε τις πολιτικές ομάδες. Και όλοι γνωρίζουμε τους συμβιβασμού ε, που πρέπει να γίνουν για να καταλήξουμε σε αυτή την κοινή θέση. Και τι γίνεται, πάνε οι συγκητές στο Συμβούλιο και βλέπουν αγγίλες. Και τι σημαίνουν οι αγγίλες. Οι αγγίλες σημαίνουν ότι αυτό δεν θα συζητηθεί. Θεωρώ πως το επόμενο κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ε, θα είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και θα πρέπει να βγουν από αυτή. Και αυτό δεν θα γίνει όταν υπάρχουν φράσεις όπως «αυτό δεν θα το συζητήσουμε». Τι σημαίνει αυτό, δεν θα το συζητήσουμε γιατί βρίσκεται σε ένα διαπραγματευτικό κουτί, ε, διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις μόνο. Τι, τι είναι όλα αυτά επαναλαμβάνω, δεν θα με εξέπλητε εάν το επόμενο κοινοβούλιο βάλει και αυτό τι δικέ του αγγείλε και πει: Ωραία, αυτέ είναι οι δικέ σα αγγείλε, αυτέ είναι οι δικέ μα, δεν θα συζητήσουμε το ένα, δεν θα συζητήσουμε το άλλο. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι όμω. Θεωρώ πω η διαπραγματευτική μα θέση, όχι τελική, θα πρέπει να είναι αρκετά σαφή και να έχουμε συμφωνήσει όλοι από κοινού προτού περάσουμε σε επόμενε διαπραγματεύσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν και οι συγητέ του Κοινοβουλίου, διότι πρέπει να γίνει σωστό συντονισμός με τους ε, συντονιστέ όλων των τομεακών πολιτικών, όλων των πολιτικών ομάδων και να είστε σίγουροι πως μετά τις ευρωεκλογέ τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν θα είναι εύκολο το Κοινοβούλιο να δεχτεί οποιαδήποτε λύση. Το θέμα δεν είναι να αντιταχθεί σε αυτές τις λύσεις, αλλά να βρεθεί μια συμβιβαστική κοινά αποδεκτή λύση. Όπως σας είπα, όπως, ε, όσο δύσκολο είναι και στο Συμβούλιο, τόσο δύσκολο είναι και εδώ. Και βλέπετε, ολοένα και συχνότερα, όπως είπε και ο, και ο Γενικός Διευθυντής στο Συμβούλιο, ότι διαβάζουν μεγάλη προσοχή τα έγγραφα και αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση του τι συνεπάγεται η κάθε λέξη. Και κάτι τελευταίο οι ευρωβουλευτές προέρχονται από ε, πολιτικά κόμματα που είναι είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Δεν μιλάμε για κάποια ε, για ανθρώπους από απομονωμένες νησίδες κάπου στη μέση του πουθενά. Μιλάμε τώρα για βουλευτές κομμάτων που κυβερνούν ή είναι στην αντιπολίτευση. Και αυτό το πολιτικό παιχνίδι περιπλέκει την κατάσταση. Αλλά το σίγουρο είναι ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο, καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο καλύτερα και είμαστε πιο πρόθυμοι να συμβαστούμε για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Δεν ε, νομίζω επίσης, ε, όπως είπε και ο συνάδελφος, πρέπει να μπλοκάρουμε το ε, πι. Αυτό δεν είναι σοβαρή απάντηση. Ούτε αφελείς είμαστε, ούτε τίποτα άλλο. Θα ξεκινήσει το νέο πολιτισμο συνομικό πλαίσιο το 2021. Θα είναι μετά τις εκλογές. Αν ήταν πριν τις εκλογές δεν θα είχε σημασία. Τώρα όμως θα ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογέ και το Κοινοβούλιο λοιπόν γνωρίζει πως θα έχει χρόνο μεταξύ 2020 και 2021 και εκεί θα γίνουν οι διάφορες πολιτικές ζημώσεις. Ευχαριστώ. Ε, φυσικά, η μεγάλη διαφορά μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου φυσικά είναι ότι καθημερινά το Κοινοβούλιο ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανησυχεί για αυτήν. Ενώ στο Συμβούλιο έχουμε κάτι υπουργού οι οποίοι πρωτίστω ασχολούνται με τι εθνικέ του υποθέσει και που ενίοτε συναντιόνται για να συζητήσουν την Ευρώπη. Και για θέματα προπολογισμού δεν συμβάλλουν και ιδιαίτερα παρότι υπάρχει πραγματικός ε, προϋπολογισμός το 1%, τα 3 τέταρτα καταλήγουν ε, με αναδιανομή στα κράτη-μέλη, μερικές φορές και με αυξήσεις. Ε. Η άλλη μεγάλη πρόκληση που θα έχει να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο αναμφίβολα θα είναι ενδεχομένω και το να διευκολύνει για να γίνει πιο συνεκτικός ο ευρωπαϊκός προπολογισμό να διευκολύνει τη μεταφορά ε, κακώς χρησιμοποιημένων δαπανών σε εθνικό επίπεδο προ τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να δείξει ότι η προσθέμενη αξία τη Ευρώπη δεν είναι ότι αυξάνει γενικά τι δημόσιε δαπάνε, αλλά ότι μεταφέρει ορισμένε δαπάνε που τα κράτη δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά για να διατηρήσουν την κυριαρχία του σε ορισμένου τομεί και ότι αυτέ οι δαπάνε μπορούν να μεταφερθούν λοιπόν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα κλείσουμε το ε, θέμα αυτό ε, του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Αλλά πιστεύω, αγαπητοί συναδέλφοι, θα πρέπει να είστε περήφανοι για το όσο έχουμε επιτύχει. Είναι αρκετά δημοκρατική διαδικασία σε τελική ανάλυση. Δεν θα ψηφιστεί πριν τις εκλογές ο προπολογισμός 2021-2027, διότι ε, και οι υποψήφοι θα πρέπει να προετοιμάσουν τις πιθανές επιλογές και όχι να πούν ε, ξέρετε ότι ψηφίστε ποιον θέλετε, αλλά ούτως ή άλλως ο προπλογισμός έχει γίνει ε, και πέραν ε, ε της ε, θητείας για την οποία εμείς είμαστε υποψήφοι. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης που προτείνεται από τον κύριο Γκάιερ. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί την καινοτομία. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο κύριος Σάνς Γκάιερ θα βρίσκεται εδώ σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε ε, τον Ωραλία Ρουμπιό από το Ίδρυμα Ζακ Ντελόρ στο Παρίσι και τον ε, Μαρκ Καπελέτσια από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής. την καινοτομία, την περιγράφει το 2010 η Κομισιόν στο καλύτερο μέσο που έχουμε για την επίλυση των προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας. Είτε πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, για την ενεργειακή ένδυα, είτε για του ολοένα και σπανιότερου πόρου, όχι ιδίους πόρου και για το πρόβλημα τη υγεία και τη γέρεση του πληθυσμού. Θα πρέπει λοιπόν η καινοτομία να τεθεί στο επίκεντρο τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Πώ αυτό μεταφράστηκε σε ευρωπαϊκέ χρηματοδοτήσει, ε, τι ε, μαθήματα που κομίσαμε για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ακούσουμε τι εμπειρογνώμονές μα Μια παρουσίαση περίπου 15 λεπτών το πολύ. Και έτσι έχουμε στη διάθεσή μας λοιπόν μισή ώρα μετά για συζήτηση. Ποιος θα ήθελε να πάρει πρώτο λόγο. Η κυρία Πιλάτη, κυρία Ρούμπιο. Κυρία Ρούμπιο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω την παρουσίαση στα αγγλικά, διότι η μελέτη έχει συνταχθεί στα αγγλικά. Η μελέτη αυτή λοιπόν έγινε από το Ινστιτούτο EPC στο Βερολίνο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής δηλαδή, και στην μελέτη θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε πόσο ο υφιστάμενος ε, προπολογισμό, το, το υφιστάμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει την κατάσταση μετά το 2020 και πώς προσεγγίζει την καινοτομία και την χρηματοδότησή της από το 2021 μέχρι το 2027 και μετά θα ε, αναφερθούμε σε κάποιες συστάσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πώς μεταφράζονται όλα αυτά. Σε πέντε διαφορετικούς στόχους. Μας ζητήθηκε να εκτιμήσουμε το, τα ποσά χρηματοδότησης ε, άμεσης ή έμεσης στην καινοτομία, να εξετάσουμε τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ε, πηγών καινοτομία, να αξιολογήσουμε τη λειτουργία και τον αντίκτυπο των εταιρικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν την καινοτομία, να ε, διερευνήσουμε το ρόλο των χρηματοοικονομικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα στηρίξουν την ε, καινοτομία και ε, να διεξαθεί μια ανάλυση ως προς την προσέγγιση στην καινοτομία για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η μελέτη λοιπόν ε, διεξήχθη μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2019 και αφού συμπεριλάμβανε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την πολιτική καινοτομία και την ίδια, και, την, ίδια την καινοτομία. Είχαμε στο πλαίσιο της έρευνας περίπου 30 συνεντεύξεις με υψηλά αισθάμενα στη λέξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ε, ΕΤΕΠ και διαφόρων άλλων ε, θεσμικών οργάνων, μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου για παράδειγμα κτλ. Είναι σημαντικό να δούμε ότι δεν υπάρχει ένας μόνο ορισμός ε, της καινοτομίας και της χρηματοδότησης της καινοτομίας. Στην εκτίμησή μας λοιπόν δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο, μία μέθοδο την οποία χρησιμοποιήσαμε για να αξιολογήσουμε τις διαφορές μορφές ε, καινοτομίας. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει έναν ορισμό βασισμένο στο εγχειρίδιο του ε, ΟΣΑ, το εγχειρίδιο Όσλο, ο ορισμό αυτό είναι αρκετά ευρύ, διότι είναι και υποκειμενικό, α μην ξεχνάμε. Η καινοτομία λοιπόν ορίζεται ω οποιαδήποτε αλλαγή που ε, συνεπάγεται κάτι καινούριο για εκείνον που το δέχεται. Υπάρχουν λοιπόν καινοτομίε ε, σε διάφορους τομείς και στους τομείς πολιτικής και στον ορισμό αυτό εμείς ε, προσθέσαμε και μία ταξινόμηση των ε, διαφόρων δράσεων στήριξης της χρηματοδότησης της ε, καινοτομίας από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αναλύσουμε τις διάφορες πτυχές της καινοτομίας εμπορική καινοτομία για παράδειγμα, διάδοση καινοτομίας, ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή γνώσεων. Είναι πολλές οι και γι' αυτό χρειάζεται και χρηματοδότηση σε πολλές κατευθύνσεις. Επίσης, άμεσες ενισχύσεις, άμεση χρηματοδότηση σε διάφορα project έρευνας και ανάπτυξης και αυτά στηρίζουν την καινοτομία. Και κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για να ε, εξετάσει τις ε, κυριότερες ε, μορφές χρηματοδότησης από τον ε, ενωσιακό προϋπολογισμό. Έχουμε κάνει κάποιες εκτιμήσεις βέβαια για τη χρηματοδότηση καινοτομίας βασισμένες στα κονδύλια που διατίθενται. Βέβαια, δεν είχαμε τον ε, κατάλληλο χρόνο για να κάνουμε εκτίμηση αντικτύπου αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά κοιτάξαμε τα κυριότερα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από τον προπολογισμό τη Ένωση, τα οποία θα επιφέρουν καινοτομία. Στην ανάλυση, λοιπόν, προέκυψαν τα εξή νούμερα. 150 δισεκατομμύρια Προ στήριξη τη καινοτομία, δηλαδή περίπου το 14% του συνολικού πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Από αυτά τα 150, τα 62 είναι από τον ε, ορίζοντα 2020, Εκτό από τον ε, προϋπολογισμό για την ε, έρευνα. 53 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 33,3 από άλλα προγράμματα. Ε, τώρα, πέρα από τον ορίζοντα 2020. Χρηματοδοτείται η καινοτομία σε άλλου τομεί, την ενέργεια, τι μεταφορέ, το κλίμα, 12,9 δισεκατομμύρια, διάστημα, 11,3 δισεκατομμύρια, ε, γεωργία και αλία, 1,7 δισεκατομμύρια, κοινωνικά ζητήματα και υγεία, 0,13 δισεκατομμύρια και ασφαλεία και άμυνα, 0,09. Περισσότερε λεπτομέρειε θα βρείτε στην ε, αναλυτική μελέτη. Έπειτα, στην επόμενη διαφάνεια. Προσπαθήσαμε να δούμε τις συνέργειες μεταξύ των ε, προγραμμάτων της Ένωσης που στηρίζουν την καινοτομία. Με βάση τους ε, στόχους που έχουν κοινού. Βρήκαμε δύο κύριες πηγές, τον ορίζοντα 2020 και το ΕΣΥΦ, ιδιαίτερα το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία έτη για την προώθηση συνεργειών που θα στηρίξουν την περιφερειακή ανάπτυξη και τη δυνατότητα των περιφερειών να συντονίσουν καλύτερα την χρηματοδότηση από αυτά τα προγράμματα με την χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα. Αυτό προέκυψε και από τις συνομιλίες που είχαμε. Βλέπουμε πως είναι ακόμα περιορισμένες οι συνέργειες για πολλούς λόγους. Ακόμα υπάρχουν ρυθμιστικά προβλήματα τα οποία ε, εμποδίζουν την ε, χρηματοδότηση Επίσης, αδυναμία στον συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων που έχουν διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο και ε, των υπολείπων. Επίσης υπάρχουν διαφορές γεωγραφικού χαρακτήρα. Ορισμένες περιφέρειες λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τον ορίζοντα 2020 για παράδειγμα και τέλος υπάρχουν οι ε, κίνδυνοι επικαλύψεων. Μετά, Κοιτάξαμε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που στηρίζουν την καινοτομία και τις κοινωνικές προκλήσεις. Εντοπίσαμε 7 κύριες κοινωνικές προκλήσεις και τις ε, συγκρίναμε με την χρηματοδότηση της Ένωσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Τώρα, δυστυχώς, δεν είχαμε χρόνο να βάλουμε όλες αυτές ε, τις ε, προκλήσεις στα, στις διαφάνειες, όμως θα τις βρείτε στη μελέτη. Τα ευρήματά μας είχαν ως εξής. Υπάρχει υπάρχουν ακόμα πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες χρηματοδότησης της καινοτομίας. Ε, για παράδειγμα, βλέπετε στον τομέα της μεταφοράς, της ενέργειας, ε, της ε, κοινωνική ασφάλεια. ασφάλειας. Μπορεί, ας πούμε, η διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη να χρηματοδοτήσει διάφορα άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται και από τον ορίζοντα 2020 ή να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά κάποια προγράμματα. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία αναφέρονται είτε ως υποσχέσεις για το μέλλον, είτε στην ε, αρχή ως απρεμία, όμως δεν έχουν υλοποιηθεί. Έπειτα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για συνδυαστικές προσπάθειες χρηματοδότησης και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τον Ιούστα 2020 για ορισμένες περιφέρειες. Εδώ βλέπουμε ότι ορισμένες περιφέρειες επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν ε, προγράμματα ε, που έχουν να κάνουν με την ευφύ εξειδίκευση. Υπάρχει κάποια προτίμηση δηλαδή εκεί. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είδαμε επικαλύψεις, ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας για την κυβερνασφάλεια. Στην περίπτωση τώρα εταιρικών σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωσης που στηρίζουν την καινοτομία. Αξιολογήσαμε τον συνολικό αντίκτυπο της εταιρικής αυτής σχέσης. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα που αναλύσαμε που ανήκουν σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες εταιρικών σχέσεων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε τα προγράμματα αυτά που χρηματοδοτούνται από την Ένωση. Υπάρχει η πλατφόρμα τεχνολογίας, η κοινή πρωτοβουλία για τεχνολογία, οι σχέσεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα, οι σχετικές συμβάσεις, μεταξύ άλλων. Όπως σας είπα, δεν είχαμε το χρόνο να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο όλων αυτών των ε, εταιρικών σχέσεων σε όλες τις ε, πλατφόρμες αυτές. Στην περίπτωση των ε, GTI και των CPPP, τα ΣΔΙΤ λοιπόν είδαμε κάποια στοιχεία του ορίζοντα 2020 που χρηματοδότησαν άμεσα τα προγράμματα αυτά και στο σύνολό τους αποτελούν το 20% της συνολικής χρηματοδότησης ε, στο πρόγραμμα ορίζοντας 2020. Αυτέ λοιπόν οι εταιρικέ σχέσει αποτελούν το 20% τη συνολική χρηματοδότηση. Τώρα, ε, μπορείτε να κοιτάξετε και εσεί την μελέτη. Προσπάθησα να κάνω μία σύνοψη και θα κάνω και μία σύνοψη των συμπερασμάτων, γιατί μέσα σε 15 λεπτά καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να τα αναφέρουμε όλα. Υπάρχουν ε, πάνω από 100 συμπράξει. Έπειτα, βλέπουμε ότι συμπεραίνουμε ότι έχουν επιτύχει εν μέρει τους στόχους τους, έχουν επιτύχει μόχλευση, έχουν επιτύχει θετικά ωφέλη, όμως υπάρχουν και κίνδυνοι διαρθρωτικού χαρακτήρα και μια που οι προκλήσεις αλλάζουν όπως αλλάζουν και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ συχνά ε, παρατηρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος μπλοκαρίσματος. Πολλές φορές δηλαδή διαθέτεις κονδύλια για ένα πρόγραμμα, αλλά μετά μπλοκάρουν γιατί προκύπτει κάποιο άλλο που είναι πιο ενδιαφέρον ας πούμε. Τώρα υπάρχει ανάγκη για αρκετές διευκρινήσει ω διευκρινήσεις ως την αποστολή της ε, χρηματοδότηση των προγραμμάτων Χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν, διευκρινήσεις για το είδος της καινοτομίας που χρηματοδοτείται και στόχος είναι φυσικά οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητες μακροπρόθεσμα. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να συνδυαστούν αυτοί οι δύο στόχοι. Έπειτα, κοιτάξαμε τα δίκτυα στήριξη των εταιρικών ε, σχέσεων. Ο στόχος χρηματοδότηση εδώ είναι η διευκόλυνση συνταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. Αλλά και να δημιουργηθεί μια κοινή ατζέντα, όμως είναι πολύ δύσκολο ακόμα να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα. Τέλος πρέπει να ενσωματώσουμε τα PPP καλύτερα στο ε, συνολικό πλαίσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση και καταλήξαμε στο εξής στα 11,2 δισεκατομμύρια προς ε, έρευνα και ανάπτυξη. Το κυριότερο ταμείο είναι το ΕΦΣΥ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που στηρίζει την, κυρίως την έρευνα και την ανάπτυξη. Συνολικά λοιπόν η αξιολόγησή μας έχει δείξει πως ε, τα προγράμματα λειτουργήσαν αρκετά καλά αν τα συγκρίνουμε με την προηγούμενη ε, περίοδο προγραμματισμού, όταν όλα ήταν καινούρια, τα ποσά ήταν ε, μεγαλύτερα και υπήρχαν πολλά καινούρια χρήματα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δημιούργησε λοιπόν καλύτερες συνέργειες, στήριξε περισσότερα προγράμματα. Βέβαια, μας ε, έδωσε και πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για τον σχεδιασμό του επόμενου προγράμματος στήριξης. για τη δημιουργία δηλαδή ενό ε, ταμείου το οποίο θα στηρίζει τις ε, καινοτόμε μικρομεσαίες κυρίως ε, επιχειρήσεις. Επίσης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας επιδέχονται βελτίωση, όπως θα σα επιβεβαιώσει και το ελεκτικό συνέδριο. Έχουμε δει ότι χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι τόσο καινοτόμες όσο θα έπρεπε. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, όμως έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις. Έπειτα, ένα ακόμα έβριμα στην μελέτη είναι ότι το 2014, το 2015 μάλλον, με την δημιουργία του ΕΤΣΕ, υπήρχαν επικαλύψεις με προηγούμενα ταμεία. Και έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διορθώσει αυτές τις επικαλύψεις του έτσα με το Ίνοφιν. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το Ίνοφιν για να χρηματοδοτήσει ε, καινοτόμες επιχειρήσεις ψηλού κινδύνου. Βέβαια, πολλά έργα έχουν συγχρηματοδοτηθεί από τα δύο ταμεία και σε αυτή την περίπτωση το Ίνοφιν παρέχει την πρώτη και την ε, τελευταία ε, δόση στήριξη. Τώρα, σε ορισμένες ε, συνεντεύξεις ε, διατυπώθηκαν αμφιβολίες για την μελλοντική ικανότητα του Ταμείου να στηρίξει την καινοτομία, διότι όπως γνωρίζετε οι εγγύησεις είναι μερικές το Ευρωπαϊκό Τομείο Στρατηγικών Επενδύσεων χρηματοδοτεί 100% προγράμματα, όπως ξέρετε, όπως και το Ινοφίν. οπότε ε, υπάρχει κάποιος κίνδυνος να μην ε, σημειωθεί επιτυχία σε ένα project. Μετά, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο περιθώριο ευελιξίας, να συνεχίσουμε με να στηρίζουμε καινοτόμε επιχειρήσει ε, υψηλού κινδύνου, όμως ε, να μην παραβλέπουμε και τις ε, επιχειρήσεις και τα έργα χαμηλού κινδύνου. Τέλος, είδαμε ότι υπάρχει έλλειψη στήριξη σε υψηλά καινοτόμε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο εξάπλωση. Στόχος λοιπόν είναι αυτό να αλλάξει, να στραφούν οι ενισχύσεις σε υψηλά καινοτόμας επιχειρήσεις. Βέβαια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζει αυτές τις υψηλά καινοτόμας επιχειρήσεις στο ξεκίνημά τους. Όμως, όταν έχουν ξεπεράσει οι επιχειρήσεις σε αυτό το στάδιο, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουν να διατηρήσουν μάλλον αυτήν την ε, ταχύτητα χωρίς πρόσθετη στήριξη. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να υπήρχε ένα χρηματοδοτικό μέσο που θα βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις και αργότερα. Τέλος, ορισμένα στοιχεία που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις μας είναι ότι οι... πολλά από τα χρηματοδοτούμενα έργα έχουν αρκετά περίπλοκο χαρακτήρα και γι' αυτό είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος. Τέλος, συστάσεις. Πριν από αυτό, να σας πω για την προσέγγιση στη χρηματοδότηση υπό το υφιστάμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε γενικές γραμμές, με μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε έργα που χαρακτηρίζονται από ψηφιακή καινοτομία, τώρα δηλαδή σε σύγκριση με το επόμενο πολιτισμο-οικονομικό πλαίσιο. Επίσης υπάρχει στήριξη σε ερηξικέλευτες ε, καινοτομίε της αγοράς. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό είναι και κινητήριο δύναμη πίσω από αυτό το Συμβούλιο Καινοτομίας. Έπειτα, δημιουργία στόχων, αποστολών, που θα εστιάσουν καλύτερα σε συγκεκριμένα έργα έρευνας και κοινοτομίας. Αν δούμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες που τον διέπουν, θα παρατηρήσουμε ότι ακόμα δεν υπάρχουν αρκετές συνέργειες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν περισσότερα προς την ε, κατεύθυνση αυτή, περισσότερες συνέργειες. Μετά περνάμε στις συστάσεις του. Έξι συστάσεις υπάρχουν στη μελέτη μας. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει μεθοδολογία καλύτερης ε, παρακολούθησης και στήριξης ε, της ε, χρηματοδότησης και Χρειάζεται λοιπόν μεθοδολογία, την οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται κάτι δύσκολο, κάτι περίπλοκο. Αλλά χρειάζεται έστω ένα πλαίσιο ε, που να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για να πούμε ότι αυτό ας πούμε ναι είναι ε, καινοτόμο, αυτό όχι. Και αυτό να εφαρμοστεί σε όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα, έτσι ώστε να εντοπίσουμε τους στόχους της καινοτομίας για να λάβουν και χρηματοδότηση τα αντίστοιχα έργα. Έπειτα, μία διαφορετική προσέγγιση προσανατολισμένη στον αντίκτυπο. Πολλέ φορέ βλέπουμε ότι τα ενωσιακά προγράμματα χρηματοδοτούν μεν την καινοτομία, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν αν η χρηματοδότηση αυτή θα αλλάξει κάτι, θα αυξήσει την καινοτομία, θα δημιουργήσει καινοτομία ή θα τη διαδώσει. Προτείνουμε λοιπόν να διασφαλίζεται ότι η χρηματοδότηση για την καινοτομία θα έχει συγκεκριμένους στόχους. Θα υπάρχει λοιπόν ένα, ε, μια, ένας κατάλογος, ένα checklist που θα λέει ποιος είναι ο στόχος, τι θέλουμε να επιτύχουμε, πού θα, ε, τι θα χρηματοδοτηθεί. Αυτό θα γίνει βέβαια και μετά από τη δημιουργία της κατάλληλης νομικής βάσης. Έπειτα, κοιτάξαμε συνολικά την ε, χρηματοδότηση και είδαμε ότι σε πολλούς τομείς πολιτικής η χρηματοδότηση δεν ήταν η κινητήριος δύναμη της ε, καινοτομίας, αλλά όπως για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, υπήρχαν συγκεκριμένοι στόχοι, ενεργειακή απόδοση, όπου ενισχύθηκαν επιχειρήσεις που είχαν αυτό το συγκεκριμένο στόχο. Προσπαθούμε λοιπόν εδώ να επικεντρωθούμε σε καινοτομίες για την ε, βελτίωση της ε, γεωργίας, για παράδειγμα. Πέντε. Σύνδεση με τον Ευρωπαϊ... των ευρωπαϊκών PPP με τις ε, αποστολές. Προσανατολισμός στον αντίκτυπο, λοιπόν. έτσι ώστε να λύσουμε το πρόβλημα αυτού του κλειδώματος των πόρων. Και τέλος, μια, ένας ε, νέος ορισμός των ε, μέσων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υφιστάμενες προκλήσεις και στα κενά που δημιουργούνται στην αγορά. Εδώ θα βοηθήσει και ο συνδυασμός ταμείων. Συνδυαστική χρηματοδότηση λοιπόν για επιχειρήσεις οι οποίες ε, τη χρειάζονται. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα αξιολογήσει αν το InvestEU θα μπορέσει να καλύψει αυτές τις ανάγκες ή αν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καινούριο ταμείο, ξεχωριστό από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Merci, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ξεκάθαρη αυτή παρουσίαση και τις πολύ ξεκάθαρες αυτές συστάσεις. Ε, χθες ψηφίσαμε το InvestEU. Δεν ξέρω αν μπορούμε να επηρεάσουμε με τις συστάσεις αυτές το InvestEU. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Γκάγερ, που είναι και αυτός ο οποίος είχε θελήσει να γίνει και αυτή η μελέτη, πώς θα μπορούσε να μας πει κάποια σχόλια. Ähm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η βασική ιδέα που είχα Όταν συζητούσαμε με άλλους ε, το πέριγραμμα αυτής της μελέτης ήταν να δούμε σε ποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματα που τα γνωρίζουμε όλοι θα μπορούσαμε να προωθήσουμε το καινοτόμο δυναμικό, να το ενισχύσουμε, μπορώ να το πω έτσι. Αν αποφασίζουμε για τα προγράμματα ε, που θέλουμε να προωθήσουμε και για τις Ευρωπαίες πολίτες πρέπει να δούμε πώς ε, προχωρούν, τι συνέχεια δίνεται, αν επιτυχάνονται οι στόχοι. Και η βασική λοιπόν ιδέα ήταν να φανεί το δυναμικό για επενδύσεις που μπορούμε να βρούμε σε προγράμματα τα οποία είναι ήδη γνωστά. Και θεωρώ ότι μας έδωσε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στοιχεία αυτή η μελέτη. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια στη επιτροπή είναι τόσο σημαντικό. Ίσως για την Ήτρε ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ε, δίνονται κάποιες ενδείξει και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι μπορεί να κάνει ώστε να είναι πιο ορατό ε, το δυναμικό αυτό ε, σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Εμεί, επειδή δεν έχουμε σχετικέ παράμετρους, δεν μπορούμε να μετρήσουμε το δυναμικό καινοτομία και αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία που νομίζω ότι μπορεί να την εκμεταλλευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εκπονήσει τέτοιου είδου παραμέτρου. Και επίση θεωρώ ότι είναι σημαντικό που δεν θα την είχαμε ε, ε, αυτή τη νέα ιδέα αλλιώς, αν δεν είχαμε ακούσει αυτή τη μελέτη, είναι τι μπορεί να γίνει για στο πλαίσιο της νομοθεσίας, όχι μόνο δηλαδή στο πεδίο της χρηματοδότησης, αν δηλαδή και στη νομοθεσία μπορούμε να βρούμε παραμέτρους για με τις οποίες θα μετρήσουμε αυτό το καινοτόμο δυναμικό. Αυτό θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ε, η καινοτομία, η γνώση και όλα αυτά πράγματι είναι σημαντικά και ε, σε ποιους τομείς κοινωνικούς ε, μπορούμε να προωθήσουμε την καινοτομία και πρέπει να ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολισμού, η κυρία Γκρέσλε μπορεί να έχει τις δικές της απόψεις. Σίγουρα μπορούμε να συζητήσουμε εκεί αλλά όχι μόνο στις δικές μας αυτές επιτροπές, αλλά και σε άλλες επιτροπές που ασχολούνται με τη διατύπωση νομοθετημάτων ή την εκπόνηση προγραμμάτων. και αν θέλουμε να πάρουμε σοβαρά τη δουλειά μας θα πρέπει να μας απασχολήσει και το τι έχουμε επιτύχει, το τι επιτυγχάνουμε τέλος πάντων με τις επενδύσεις μας. Αν σκεφτεί κανείς ε, την καινοτομία, μπορεί να είναι μια επένδυση πράγματι ε, τόσο σημαντική, να προωθεί τόσο πολύ την καινοτομία όσο νομίζαμε. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να τα μελετήσουμε. Νομίζω ότι μας δώσατε με τη μελέτη σας πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που θα μας παρακινήσουν και θα είναι ένα κίνητρο για να αξιοποιήσουμε τα πορίσματα. και τις, ε, τα PPP, τα SDIT ε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να το μελετήσουμε και νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ καλή ε, και σε αυτό το πεδίο η μελέτη σας γιατί περιλαμβάνει πολλές ιδέες που είναι σημαντικές για τη δική μου πολιτική εργασία και νομίζω ότι χρήζουν περαιτέρω συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο η κυρία Μάλιτιτ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πολύ καλή αυτή μελέτη, πλήρη μελέτη. Δύο πορίσματα θεωρώ σημαντικά. Αυτά που είναι στη διαφάνεια 10. Γιατί υπάρχει έλλειψη συντονισμού με προγράμματα σε εθνικό επίπεδο, ένα και δύο, οι αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι δυνατόν να διατηρηθεί, να αυξηθεί η υποστήριξη σε επενδύσεις ψηλού κινδύνου. Είμαστε πίσω στην Ευρώπη, νομίζω, σε ό,τι αφορά την Κίνα ή τη ΣΥΠΑ, σε επενδύσεις ε, που προωθούν την καινοτομία. Και αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Και τι πρέπει να γίνει για να στηριχθούν επενδύσεις, όχι υψηλού κινδύνου μόνο, αλλά να υποστηριχθούν και έγκαιρα και γρήγορα οι καινοτομίες αυτές. Και οι καινοτόμες επιχειρήσεις που είναι στη φάση της επέκτασης, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές νοφείς επιχειρήσεις μεν, υπάρχει όμως ένα τεράστιο πρόβλημα αναπροσαρμογής και αναβάθμισης, δηλαδή υπάρχει αυτή η νοοτροπία αναβάθμισης και αναπροσαρμογής τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάουερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση πλήρης και μπορεί να μας βοηθήσει για την μελλοντική κατάρρευση του προπολογισμού. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα την αξιοποιήσει το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προκύψει από την επόμενη θητεία και ίσως εγώ ή κανένας από τον Ηνωμένο Βασίλειο να μην είμαστε εδώ βέβαια. Ε, κάτι που τουλάχιστον γι' αυτό είναι σαφή η Βρετανική κυβέρνηση, αν και νομίζω θα μπορούσε να το έχει κάνει λίγο νωρίτερα στην πραγματεύση, είναι ότι επιθυμεί έτσι λέει ξεκάθαρα τουλάχιστον, να συνδεθεί, να παραμείνει σαδεμένη με το πρόγραμμα Horizon 2020. Άρα ο προπολογισμό εδώ θα είναι πιο σημαντικός από ό,τι θα ήταν. Αλλιώ βέβαια θα δούμε την τελική έκβαση. Καλό νομίζω να φέρουμε ήδη από τώρα. Δύο τομείς ε, πιο πολύ με μουσική προσοχή. Το πρώτο είναι το επίπεδο του ΕΤΠΑ και πώς συνεισφέρει στην καινοτομία. Με βάση εκτιμήσεις έκθεσης, αυτό το ποσοστό νομίζω το 7% ήταν πολύ μεγαλύτερο στην πράξη. Επίσης, περιφέρει και πολιτική και υποστήριξη των επενδύσεων της καινοτομίας θα πρέπει να μας απασχολήσει εκ του σύνεγγις το θέμα. Πρέπει να είναι ευφυεί οι ε, επενδύσει και στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μια ευφυή, βιώσιμη, πολύ πιο βιώσιμη ιδέα από άλλε παραδοσιακέ επενδύσει. Για τι υποδομέ. που δεν πάντα βιώσιμη σε επενδύσει που κάνουμε εκεί και γιατί να ενισχύουμε ε, τις υποδομές ε, στις μετακινήσεις εάν δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθούμε ίσως. Τέλος πάντων. Και η κυρία Μάλετιτς έθιξε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δηλαδή είμαστε καλοί στην καινοτομία και στην έρευνα στην Ευρώπη, αλλά δεν είμαστε πάντα τόσο καλοί στο να την αξιοποιούμε και να την εκμεταλλευόμαστε την ε, καινοτομία και την έρευνα. Είδαμε και τα δύο-τρία χρόνια τι γίνεται με την επέκταση του κλάδου του επιχειρηματικού κινδύνου. Είναι υπανάπτυκτη σε σχέση με το αντίστοιχο τον ήπα; Ή αντίστοιχη ε, με την Κίνα που είναι κρατικές επενδύσεις εκεί. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην Ευρώπη. Είναι μια μείζον πρόκληση. Και πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσει αυτέ δεν θα οδηγήσουν απλά και μόνο σε μια κατάσταση που θα έχουμε δημόσιε επενδύσει μέσω τη Ένωση και των Εθνικών Ταμείων με ιδιωτικοποίηση των κερδών λόγω του χειπηρηματικού κινδύνου. και του κεφάλαιου επιχειρηματικού κινδύνου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ανακυκλώσουμε μερικά από αυτά που στη μελλοντική έρευνα. Είναι μια από τι προκλήσει. Ελπίζω να συνεχιστεί λοιπόν αυτό το έργο. Και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα συζήτηση μέσω του οποίου να εξετάσουμε τον προεπολισμό διαφορετικό μάτι με γνώμονα την καινοτομία, ίσω θα μπορούσαμε να είχαμε μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία νωρί στην επόμενη θητεία να ευχαριστήσω τους ε, συντάξεις και τον Γένς για την ενδιαφέρουσα αυτή πρόταση που είχε. Merci. Ευχαριστούμε, κύριο Άλμπρεχτ. Ε, ναι, ε, βάσει των όσων είπαν οι προλαλήσαντες, να δώσω κι εγώ μια άλλη οπτική γωνία. Το θέμα δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφέρειας Ανάπτυξης και η Πολιτική Συνοχής ε, και οι σχετικές καινοτομίες. Αυτά που αναφέρατε εδώ είναι πολύ σημαντικά αυτό που είναι σημαντικό είναι η συνέργεια μεταξύ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ε, καινοτομία ε, και περιφερειακής ανάπτυξης. Και αυτό υπόθηκε μόλις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το αποτέλεσμα, την έρευνα που πραγματοποιούμε εκεί. Και αληθεύει αυτό η συνέργεια, για παράδειγμα, μεταξύ του ορίζοντα 2020 ε, και των άλλων είναι περιορισμένη. Για ποιο λόγο, διότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Από τη μια έχουμε το Horizon 2020, έρευνα κτλ. Και τα υπόλοιπα αφορούν τον πραγματικό κόσμο, πρακτικά ε, προγράμματα και προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι αυτά είναι καινοτόμα ενώ ταυτόχρονα ε, κάνουμε την έρευνα για να κάνουμε πιο καινοτόμα τα προγράμματα αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι από τα βασικά στοιχεία ότι χρειάζεται συνέργεια μεταξύ διαφορετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι περίπλοκο. Πρόκειται για διαφορετικές διευθύνσεις, ε, ε, διαφορετικούς επιτρόπους κτλ. Αλλά η τάση σήμερα, αν δει κανείς την πολιτική συνοχή, συνοχής, είναι να παίρνει ένα χρήματα από την πολιτική συνοχή και να τα μεταφέρεις σε άλλα προγράμματα και μετά να κάνει τη συνέργεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ήθελα να το υπογραμμίσω αυτή τη διάσταση που θεωρώ σημαντική. Ευχαριστώ. Merci, je vois pas δεν βλέπω να ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Ευχαριστούμε. Να πω δύο λόγια και εγώ. Εγώ ήρθα σε επαφή με του υπευθύνου μια καινοτόμου μικρομεσαίας επιχείρηση και ήθελα να υποφεληθούν από μια επιχορήγηση 50.000 ευρώ για καινοτομία. Όπω προβλέπετε και του είδα. Δεν ήξεραν τι να κάνουν Ε, είχαν ε, βαθμολογία τέτοια, αξιολόγηση τέτοια που ήταν πολύ κοντά σε αυτήν για να μπορεί να πάρει κανείς επιχορήγηση και μετά ακολούθησε απογοήτευση. Αναρωτιέμαι δηλαδή κατά πόσο οι αυστηρέ διαδικασίε που έχουμε, οι οποίε μερικέ φορέ είναι και αυθαίρετε, γιατί αφού δεν έχουμε αρκετέ πιστώσει, ε, συχνά δίνουμε αξιολογήσει, κάτι περίπλοκο και κάποιο βρίσκεται ακριβώ πάνω από την αξιολόγηση, ακριβώ κάτω από το κατόφλι, σα φαίνεται σωστή. Αυτή η αξιολόγηση κυρίες και κύριοι και μετά τελικά όλοι αυτοί οι κανονισμοί στους οποίους συμμετέχουμε και εμείς ε, συνάδουν με την έννοια της καινοτομίας σε τελική ανάλυση. Μήπω τελικά είναι υπερβολικά περίπλοκα όλα αυτά, ή μήπως είναι υπερβολικά πολλές οι για να συζητάμε περί καινοτομίας. Πώ να υπάρξει πειραματισμό όταν έχουν προβλεφθεί όλα εκ των προτέρων. Εκεί έχουμε μια ευρωπαϊκή αντίφαση. Και τέλο, ε, αν πάτε να δείτε του μηχανισμού που υπάρχουν παγκοσμίω, Κίνα, ΗΠΑ, οι δικέ του δημόσιε κρατικέ ε, προσεγγίσει μήπω είναι πιο λογικέ, πιο αποτελεσματικέ, πιο φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Αγαπητή κυρία, έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε στι διάφορε ερωτήσει. <laughs> Well, I um, just two or three comments on what has been said. Δύο λόγια θέλω να πω σε αυτά που άκουσα. Τώρα συμφωνώ απόλυτα για την καινοτομία υψηλού κινδύνου. Θα διαφέρει βέβαια το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο από το υφιστάμενο, διότι διαφέρει και το συγκείμενο Ορισμό τη ε, καινοτομία. Τώρα είμαστε στη μέση τη κρίση. Ξεκίνησα με το προηγούμενο πολιτισμό συνομικό πλαίσιο του 2014 και τότε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ο όγκο ε, τη ε, χρηματοδότηση ήταν μεγαλύτερο. Φυσικά στηρίχθηκαν πολλά περισσότερα έργα, όμω εκείνα που πλήγησαν περισσότερο από την κρίση ήταν αυτά που είχαν χαρακτήρα καινοτομία υψηλού κινδύνου. Τώρα, αν δείτε την έκθεση της ΕΤΕΠ, την ετήσια έκθεση της ΕΤΕΠ, θα δείτε ότι δεν είναι όλες οι καινοτόμες επιχειρήσεις υπό τέτοια πίεση. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις ε, καινοτομία οι οποίες ε, ονομάζονται adapters. Προσαρμόζονται δηλαδή στα ε, δεδομένα, γίνονται πιο εμπορικές, συνδυάζουν την ε, καινοτομία με τον εμπορικό χαρακτήρα. Αυτό είναι ε, νέος ε, τύπος επιχείρησης. Έτσι λοιπόν δεν υφίστανται περιορισμούς. Αν συνεχίσουμε λοιπόν να στηρίζουμε, να χρηματοδοτούμε τις επιχειρήσεις αυτές, θα είναι κατάλληλο ή θα πρέπει να εστιάσει η θα πρεπει να εστιασει χρηματοδοτηση σε καινοτομία Υψηλή εξειδίκευση, κάτι που μπορεί να στηρίξει μετά και η αγορά. Εδώ υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζει αρκετά αυτού του είδους τις επιχειρήσεις και θεωρώ πως θα έπρεπε να στηρίζονται περισσότερο οι εξικέλευτες ε, καινοτόμες επιχειρήσεις. Χρειάζεται βέβαια μια ισορροπία. Γι' αυτό πρέπει να ε, υπάρχει συμπληρωματικότητα με το εθνικό επίπεδο και να δοθεί έμφαση σε ε, χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις μεγαλύτερες από τις άλλες ή που ο ιδιωτικός τομέας δεν στηρίζει αρκετά την κοινοτομία. Τώρα, για τα χρηματοδοτικά μέσα νομίζω πως ε, θα πρέπει να προβληματιστούμε και σας καλώ να το κάνετε. Και για το scaling up. Φαίνεται πως ε, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις σχετικές ε, αναφορές και εκθέσεις. Ε, υπάρχουν προβλήματα με το επιχειρηματικό κεφάλαιο και εδώ έχουν γίνει πολλά για να βελτιωθεί η κατάσταση, όμως ακόμα υστερούμε αν συγκρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένε Πολιτείες ή με την Κίνα. Κάτι θετικό θα έλεγα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι πως έχουν καταβληθεί προσπάθειες για βελτίωση της ε, συνδυαστικής χρηματοδότησης με τις Εθνικές ε, Τράπεζες Πρόθεσης. Φυσικά υπάρχουν διαφορές στις κεφαλαίες Δεν έχουμε μία ενιαία κεφαλαία αγορά που θα ήταν καλό πιστεύω. Τώρα, συνέργειες με τον ορίζοντα 2020 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Από τη μελέτη προκύπτει ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Υπάρχει διαφορά ως προς την αντίληψη ε, του τι σημαίνει συνέργεια. Αν ας πούμε μιλήσετε με την ΓΔ ή τη ΓΔ Research θα δείτε πως υπάρχουν διαφορές. Και οι συνέργειες γίνονται αντιληπτές ως μια συνέχεια του ορίζοντα 2020. Αυτό κατά την άποψη της ΓΔ Ρίτζιο. Φυσικά έχουν ένα δίκιο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ανταποδοτικός χαρακτήρας, όμως αν χωρίσουμε τελείως τη χρηματοδότηση από τις περιφερειακές προτεραιότητες, τότε θα περιοριστούμε πάρα πολύ και θα δυσκολευτούμε στην επίτευξη συνεργειών. Σίγουρα υπάρχει ένα όριο σε αυτές τις συνέργειες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τελείως διαφορετικά μεταξύ τους προγράμματα, όμως οι συνέργειες, όπως λέει και η Γαμαδελταρίτζιο, δεν θα πρέπει να είναι μονόπλευρες, θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουν περιοχές που έχουν πρόβλημα πρόσβαση στα προγράμματα του ορίζοντα 2020. Τέλος, αυτή η αγανάκτηση από πλευρά επιχειρήσεων που δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση. Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία σχεδόν πιάνουν τα επίπεδα επιλεξιμότητας. Θα πρέπει λοιπόν να τα βοηθήσουμε έτσι ώστε να βρουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπήρξαν προβλήματα κυρίως ε, λόγω του διαφορετικού σκεπτικού, της διαφορετικής αντίληψης αν θέλετε από την εκάστοτε επιχείρηση. υπάρχουν ορισμένες επιχειρήσεις που για λίγο έχασαν χρηματοδότηση και αυτές τι επιχειρήσεις θα πρέπει να τις βοηθήσουμε βρίσκοντά τους άλλου πόρου. πόρους. Οσγκάιερ, έχετε κάποια παρατήρηση με βάση αυτά που ακούσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε, για την ε, μελέτη που παρουσιάσατε, η οποία σίγουρα θα εμπνεύσει τους ε, εισηγητές ε, για το InvestEU. Κύριε Φερνάντες. Πολύ ωραία. Θα περάσουμε λοιπόν ε, στις ψηφοφορίες. Και πριν ψηφίσουμε, προτείνω να κάνουμε μία δοκιμή. Έχετε βάλει τις κάρτες σας στις ηλεκτρονικές συσκευές. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Όχι. Κύριε Ντεπρέ, δύο κύριε Κερμαν και εγώ δεν έχουμε την κάρτα μα. Εγώ ψήφισα υπέρα, κύριε Κονμέν. Επίση. Très bien. Πολύ ωραία, μπράβο. Ε, έχουμε δύο ψήφους λοιπόν, επιπλέον. la décision de ce vote est Θετική έκβαση της ψηφοφορίας λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο ε, ψήφους ε, φυσικά οι οποίες είναι ευπρόσδεκτες. Λοιπόν το πρώτο πράγμα που θα ψηφίσουμε με οδηγεί να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με την γραπτή διαδικασία και την απόφαση των συντονιστών η γνωμοδότηση που σχετίζεται με την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΤΕΠ η επιπρόθεση νομοθετικής του Συμβουλίου για να ληφθεί υπόψη η αύξηση του κεφαλαίου ε, που θα καταβάλει η Πολωνία και η Ρουμανία. Αυτή η γνωμοδότηση παρουσιάζεται με την απλοποιημένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες βάσει του άρθρου 51. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα ψηφίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση και θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται μετά από την παρούσα συζήτηση, εφόσον φυσικά αν υπάρχει ένσταση. Ίσως η κυρία Καρδιά Ζαπάλ που συνέταξε τη γνωμοδότηση αυτή να θέλει να μας πει κάτι για τη γνωμοδότηση αυτήν. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται πράγματι για μια διαδικασία όχι απλά απλουστευμένη, αλλά και απλή, διότι με την ε, υποτιθέμενη αναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου τροποποιήθηκε το σχετικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ως ήθιστε ζητήσαμε παρά την αποχώρηση αυτή να προσπαθήσουμε να που καταστήσουμε το κεφάλαιο του Ηνωμένου Βασιλείου με νέο κεφάλαιο το οποίο θα το καταθέσουν άλλες χώρες. Αυτό βέβαια είναι ένα μικρό πρώτο βήμα. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση αυξάνεται η συμμετοχή της Πολωνίας και της Ρουμανίας γιατί ουσιαστικά όταν προσχώρησαν οι δύο αυτές χώρες ε, ε, κάλυψαν με ένα πολύ μικρό ε, ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ στο απαιτούμενο κεφάλαιο. Έχουν βιώσει με σημαντική αύξηση του ΑΕΠ όμως στο μεσοδιάστημα αυτές οι δύο χώρες και γι' αυτό μεταλλευόμαστε τα περιθώρια αυτά για να αυξήσουμε τη συμμετοχή τους. Θεωρούσα ότι είναι σημαντικό και από διαδικαστικής πλευράς πληκτιστεί τη γνωμοδότησή μας, αλλά και κυρίως γιατί με την ευκαιρία αυτή μπορούμε να πούμε ότι αν τελικά γίνει πραγματικότητα το Brexit, τα, τα κράτη-μέλη, ετέπτες θα πρέπει να καλύψουν το κεφάλαιο που θα χαθεί λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να συνεχίσουμε να ε, διατηρούμε σε ένα υψηλό επίπεδο τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε να πει κάτι για αυτή την γνωμοδότηση τη κυρία Γκαρδία Ζαμπάλ. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση. Υπάρχει αντίρρηση, ένσταση για τη γνωμοδότηση αυτή. Όχι. Οπότε θα θεωρήσουμε ότι εγκρίθηκε. Και συγχαίρω την εισηγητρία. Δεν έχουμε μεταφορές για το τμήμα 3 του προπολογισμού 2019, οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Ρίμπιχ για τις αιτήσει μεταφορά ε, που προτείνονται για τα υπόλοιπα τμήματα. Τέσσερι μεταφορές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο πρώτος ε, τομέας έχει να κάνει με το Κοινοβούλιο λοιπόν. Υπάρχει η μεταφορά C3 και θα γυρίσω στα αγγλικά. Λοιπόν, η μεταφορά αυτή έχει στόχο να μετακινήσει 100.000 ευρώ από το σημείο 3.200 απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης δηλαδή στο 16-12, μάθηση και ανάπτυξη για διάφορα project χρηματοοικονομικής διαχείρισης που χρειάζονται διοργάνωση λοιπόν. Είμαι υπέρ αυτής της μεταφοράς και μετά περνάμε στην μεταφορά C4 για ε, μεταφορά στο σημείο 3042 συνεδριάσεις, ε, ημερίδες, συνέδρια και αντιπροσωπείες με τρίτες χώρες. Πρόκειται για μεταφορά 400.000 ευρώ. Επίσης, από το σημείο 3042 η μεταφορά θα γίνει στο σημείο 3230 ε, στήριξη δημοκρατίας και οικοδόμηση ικανοτήτων για τα κοινοβούλια τρίτων χωρών και στο σημείο 3200 απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης. Περνάμε στο C5. Έχει να κάνει με την ημερομηνία αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως για παράδειγμα ε, το σημείο 1, μισθή, 1,7 εκατομμύρια ευρώ, ε, οδηπορικά έξοδα, 130.000, γενικά έξοδα 900.000, οργάνωση ε, ομάδων επισκεπτών, σχετικές δαπάνες 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι πιστώσεις θα προέλθουν από τα ε, προσωρινά κονδύλια σύμφωνα με το άρθρο 50 του εσωτερικού κανονισμού και περνάμε στο C6. Πρόκειται για μεταφορά 100.000 ευρώ ε, από αποζημιώσεις προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί που έχουν τώρα δικαίωμα λήψης αποζημίωσης για το έτος 2019. Πρόκειται λοιπόν για τη συντάξη προσωπικού με άλλα λόγια και επίσης είμαι υπέρ αυτής της μεταφορά. Αυτά κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και ε, χαρά τα να ακούσω σχόλια. Πάμε στους σκιώδες συζητητές, έχετε παρατηρήσει. Δεν βλέπω κάποιο να θέλει το λόγο. Πέραν των ε, σκιωδών, ήθελε κάποιος να πει κάτι, όχι. Ωραία, κύριε Ρούμπιγκ, λοιπόν σε 3, σε 4 και σε 6 δεν χρειάζονται ψηφοφορία, εγκρίνονται. Αντιθέτως το C5 απαιτεί ψηφοφορία. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το Πέρα ψηφοφορία. 19 υπέρ, 1 κατά και 2 τον κύριο Κολμέλ και Ντεπρέ. Ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Μόνικα Χολμάιερ, δεν έχετε ζητήσει ψηφοφορία για το ζήτημα της κτηριακής πολιτικής. Αντιθέτως, έχετε να μας προσθέσετε κάποιο σχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ε, την ε, ανανέωση του ενοικιαστηρίου για κάποια κτίρια και σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο. Για το κτίριο MO34, ανανέωση του νοικιστηρίου είναι για δύο ε, περισσότερα έτη. Το θέμα έχει προκύψει από τους ιδιοκτήτες ε, του κτηρίου, γι' αυτό λοιπόν εσείς έχετε τον λόγο. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης ε, του κτηρίου μη όμικρον 34, αν είναι επιχείρηση πίσω από την οποία κρύβονται άλλοι. Το τέλος λοιπόν του συμβολέου είναι τέλος Ιουνίου 2020. Συνολική επιφάνεια είναι 2.582 τετραγωνικά μέτρα και κάποια τετραγωνικά μέτρα ε, με αρχεία. Στο πλαίσιο λοιπόν ε, του συνολικού, της συνολικής προσπάθειας να γίνουμε πιο αποδοτική, πιο οικονομική στα κτίρια. Προσπαθούμε να βρούμε μια καινούργια λύση για το πρόβλημα αυτό. Θα σας ενημερώσω λοιπόν σχετικά με τις εξελίξεις. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι για μια διετή παράταση του ενοικιαστηρίου. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε εγκαίρω να λάβουμε όλα τα σχετικά ε, στοιχεία και πληροφορίες για να μπορέσουμε να λάβουμε μια απόφαση. Αυτά από μένα προ το παρόν. Δεν έχω άλλη να σας πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Συγητρία. Οι σκιώδει έχουν να πούν κάτι. Κύριε Χοφμάν, όχι. Κολμέλ, ούτε. πρέπει ούτε. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να εκφραστεί για αυτή την ανακοίνωση της κυρίας Χολμάιερ, κανένας. Θα κλείσουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή και θα σταματήσουμε μέχρι τις 11 και 4. Στις 11 και 4 θα έχουμε την κοινή συνεδρίαση με την ΚΟΝΤ, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Διακόπτη συνεδρίαση.